πρακτικό τη παρούς συνεδρίασης και αν δεν έχετε αντιρρήσει θα θεωρηθεί ο κατάλογος αυτός ε, γκριθής. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα υπογράψω ένα νομοθετήματα στη συναπόφαση με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού. Επίσης το πακέτο των τηλεπικοινωνιών πρέπει να σας πω θα υπογραφεί στο ημικύκλιο ε, στις 3.